τα κείμενα τα οποία ενεκρίθηκαν στη οι ολομέλειας του Μαρτίου έχουν διανεμηθεί, υπάρχουν αντίρρησεις σε σχέση με αυτά και τα πρακτικά. Εάν όχι, συνεχίζουμε.